Ε, συμφωνία Βάση του κανονισμού 69 παράγραφος 1. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έκθεση Σβόμπαντα, ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάλι έκθεση σβόμποντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μέλο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Έκθεση Βίλμετ. Θα δώσω το λόγο στους δύο συγητές, τον κύριο Βίλμοτ καταρχήν και τον κύριο Λίζε στη συνέχεια. Στην κυρία Βίλμοτ. Αυτή είναι δεύτερη ανάγνωση και αυτή η συμφωνία Πήρε πέντε χρόνια να φτάσει σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι λοιπόν που έχω μια πλατιά υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Είναι σημαντικό. Είναι... Ψηφίσουμε λοιπόν κάτι το οποίο βελτιώνει τα δικαιώματα των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ντροπή σε όλους όσους αρνούνται να το κάνουν και το καταψηφίζουν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βίλμοντ. Ο κύριος Λίζε έχει το λόγο. Παρακαλώ το μικρόφωνο. Ωραία λοιπόν. Ίσως μια σύντομη τοποθέτηση για την ε, ψηφοφορία, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Συνήθως στην συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Αλλά τώρα το UKIP ε, έκανε μια, ε, το έβαλε μια αρνητική τροπολογία και του είμαι ε, ευγνώμων γιατί μετά τη συζήτηση για το Brexit έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε πόσο συσπηρωμένο είναι το σώμα κατά των ιδεών του UKIP. Είμαστε κατά και αποφασίζουμε κάτι το οποίο είναι υπέρ της εσωτερικής αγοράς, το οποίο βελτιώνει την κατάσταση και το πίπεδο προστασία των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη και χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ε, και σε συνεργασία με την ε, Κομισιόν. Αλλά θα ήθελα να εξάρω με την ευκαιρία αυτή και όλους τους συνεργάτες που έφτασαν σε αυτό το, που συνέβαλαν στην αίσια έκβαση. Παρακαλώ λοιπόν να καταψηφίσετε την τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ελίζε. Τώρα ψηφίζουμε για την ε, πρόταση για την ε, καταψήφιση της ε, τροπολογίας. Άρχεται η τροπολογία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες, άρα εγκρίνεται και ολοκληρώνεται εδώ η δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Τώρα θα έρθουμε στην έκθεση Λίζε Καταρχήν θα ψηφίσουμε για μια επιτροπή της απόρριψης της τοποθέτησης του Συμβουλίου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και εδώ δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες, άρα λοιπόν εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Η δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται. Και φτάνουμε στην έκθεση Jill. Καταρχήν υπάρχει ε, η πρόταση να, αρνηθ, να απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, η ψηφοφορία γίνεται ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμφωνία την προσωρινή συμφωνία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση Γέσε και εδώ θα ψηφίσουμε για μια προσωρινή συμφωνία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα ολοκληρώνεται την πρώτη ανάγνωση και θα έρθουμε στην έκθεση Όλμπριχτ. Ε, ε, ονομαστική κλίση. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται μία άλλη έκθεση Olbricht. Έχουμε τις τροπολογίες 1 και 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται ε, το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Όλμπριχτ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα έρθουμε στην έκθεση Ashworth. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 33 ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 14 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Ψήφισαν άπαντες. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Για τον κανονισμό. Διαδικαστικό, συγγνώμη. Ε, πέμπτο τμήμα. Ο συνάδελφος κύριος Ρούμπιχ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω το 37.1 έχει απορριφθεί. Εδώ πρόκειται για το publishing και το general allowance. Γι' αυτό πιστεύω ότι το 5 καταπίπτει κατά συνέπεια. Κύριε Ρούμπιχ, έχω την εντύπωση ότι δεν καταπίπτει. Η παράγραφος 1 έχει γίνει δεκτή. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκτά και τα τέσσερα τμήματα. Η τροπολογία υπαριθμών 1 των Πρασίνων έχει απορριφθεί και κατά συνέπεια πήγαμε στην 9-17 και το αρχικό κείμενο. Και τα πρώτα τέσσερα τμήματα εγκρίθηκαν και τώρα ψηφίζουμε για το πέμπτο τμήμα. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 μετά την παράγραφο 17. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 παράγραφος, αρχικό κείμενο, υπέρ κατά. Αποχές, νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Εκ, 36 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 στο αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται 19 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας απορρίπτεται 23 επίσημα ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ. 28. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Εποχέ απορρίπτεται. 12 ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 40. Επίσημα ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 58 του αρχικού κειμένου ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 2 και 13 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση Γκάιερ με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Νεγκρέσκου έκθεση. Με ονομαστική κλίση είναι αναγκαία ειδική πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Φερνάντες, με ονομαστική κλίση, επίσης απαιτείται ειδική πλειοψηφία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Μωράες. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σαργεντίνη. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντας πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τεχόφσκι με ονομαστική κλίση. Ε, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της Εγκρίνεται. έκθεση Ιωσμένοβα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έκθεση Γκραπίνη με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Βάση για το γενετικά μεταλλαγμένο ε, καλαμπόκι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είναι έκθεση συναδέλφου Βαλενσιάνο και Διάθετε μέρα. Ε, παράγραφος 23, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 59. Ε, αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του έτσι όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση που εξοικονομήσαμε θα πρέπει να την τιμήσουμε ε, τάχιστα την αίθουσα εφόσον δεν θέλετε να ακούσετε τις επεξηγήσεις ψήφου και κυρίως να μην ε, παραμείνετε στους ε, διαδρόμους ε, συζητώντας. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους και ονομαστικά να τερματίσουν αυτές τις συζητήσεις.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 Ο συνάδελφος Γκραφ Λάμστορφ. Κύριε Κράμερ. Κύριε Κράμερ. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Kollege Graf Lambsdorff. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Kollege Lambsdorff. frau kollegin